κατά νότατο όριο σύμφωνα με το άρθρο 135 του κανονισμού. Το επόμενο σημείο στη σχετική ημερήσια διάταξη αφορά στους νόμους περί βλασφημίας στο Πακιστάν και δίνω το λόγο στους συντάκτες με τη σειρά για ένα λεπτό ο κύριος Τάνοκ. Κύριε Πρόεδρε, ε, οι νόμοι περιπλασιμίας στο Πακιστάν ε, προβλέπουν ε, ισόβια ή και θάνατο σε όποιον προσβάλλει το Ισλάμ. Έτσι έχουν στοχευτεί μειονότητες κατά τρόπο δυσανάλογο και ειδικά ε, Μουσουλμάνοι, Αμαδίρ, Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί και Ινδουιστές. Συχνά είναι επινοημένες οι κατηγορίες και τα πρωτοβάθμια δικαστήρια καταδικάζουν σε θάνατο. Και παρά το ότι ομολογουμένως το Πακιστάν δεν έχει εκτελέσει κανέναν για σημεία αλλά συχνά υπάρχουν άπειλες, αλλά και συχνά ε, λιντσαρίσματα και οχλοκρατία. Βεβαίως ε, παραμένει η βασική υποτίθεται προτεραιότητα του Πακιστάν ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει όμως να ενθαρρύνουμε τις ε, κυβερνήσεις να τηρήσουν το πρόγραμμα, το και το Σύνταγμα του Πακιστάν ε, δίνοντας ίσα δικαιώματα σε όλους τους πολίτες, ειδικά τις μειονότητες, γυναίκες και παιδιά. Γι' αυτό το, ε, η ομάδα μας ε, ζητά από το Πακιστάν ανάκληση αυτών των νόμων που μόνο φόβο προκαλούν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην ε, ομιλία του, στη συντακτική συνεδρίαση το Κοινοβουλίου του Πακιστάν ε, το 1947 ο Αλή Σινάπο, ιδρυτικός πατέρας ε, της κράτους του Πακιστάν ε, δήλωσε ότι οι Πακιστανοί θα έπρεπε να είναι ελεύθεροι να πηγαίνουν στα τζαμιά ή στους ναούς οποιασδήποτε άλλες θρησκείες και θα μπορούσαν να, να ανήκουν σε οποιαδήποτε θρησκεία και ή κάστα και η πίστη τους δεν θα έπρεπε να, να, έχει καμία σχέση με την ε, θέση του στο κράτος. Σάμα Μπίμπι Σαχμπάς Μασίς και ένας Ροάλ είναι τα τελευταία μόνο θύματα της, ε, της νομοθεσίας του Πακιστάν. Κάθε επεισόδιο υποτιθέμενης βλασφημίας ε, σχηματίζει μια λυσίδα αδικίας και η η συχνότητα αυξάνεται σε κάθε βήμα. Ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει το κύρος της ώστε να επιβάλλει στο Πακιστάν ε, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω των διεθνών συμβάσεων τις οποίες έχει κυρώσει και μέσα του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων. Έχει ο κύριος Βάιντεν Χόλτσερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σημαντικός εταίρος το Πακιστάν για την Ευρώπη. Γιατί? Είναι κρίμα να ακούμε πως δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πάντα έχουμε ανησυχητικά γεγονότα. Ειδικά μας ανησυχούν οι νόμοι αυτοί περί βλασιμίες. Πολιετής ποινές ε, φυλάξει, ακόμα και καταδίκες σε θάνατο για ανθρώπους που υποτίθεται ότι προσέβαλαν το Ισλάμ. Δεν είναι δυνατόν να να παραβιάζεται συστηματικά το δικαίωμα της ελεύθερης άσκησης ε, της ε, θρησκείας ε, στο Πακιστάν. Κυρίως πρέπει να υπενθυμίσουμε στο Πακιστάν πως πρέπει να σταματήσουν τα περιστατικά αυτοδικίας. Δεν χρειάζεται οχλοκρατία αλλά κράτος δικαίου. Δεν βλέπω στην αίθουσα την κυρία Τσαρανσόβα, γι' αυτό δίνω το λόγο στην κυρία Βερζιά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο πολιτικός σχετικισμός Όλο και περισσότερο πρετανεύει στο Κοινοβουλίο δυστυχώ. Ναι, εδώ πέρα έχουμε δυσμενεί διακρίσει στο Πακιστάν, αλλά ε, αυτό ε, δεν αφορά μόνο τι τις γυναίκε. Ε, Σουνίτε και, και, ε, και κόντρα στην θρησκευτική ανεκτικότητα. Πρόκειται ε, για αυτόν του νόμου για την βλασφημία. Και οπότε διώκονται, εκφοβίζονται τα πρόσωπα κακοποιούνται. Θα πρέπει επομένω όχι να γίνει αναθεώρηση όπω λέει το κείμενο, θα πρέπει να καταργηθούν αυτοί οι νόμοι, να σταματήσει αυτή η βία. Θα πρέπει να έχουμε ε, κατάργηση τη θανατική ποινή και να υπάρχει διαχωρισμό εκκλησία και κράτου. Θρησκεία και κράτου. Γι' αυτό είναι κάτι το αφόρητο. αυτά χρησιμοποιούνται για πολιτικέ σκοπιμότητε, για από κάποιους ε, ε, φονταμεταλιστές. Αυτοί θέλουν την Σαρία. Για μας δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων αυτό το κείμενο, γι' αυτό και εμείς θα το καταψηφίσουμε. Στο μεταξύ ήρθε και η κυρία Τσαρανσόβα, οπότε της δίνω το λόγο. Mr. Πρόεδρε, Ούτε ένα χρόνο δεν έχει περάσει από τότε που ψήφισαμε το τελευταίο ψήφισμα για αυτό το θέμα. Και πάλι ασχολούμαστε με την τραγωδία ε, αυτή. Ε, το Πακιστάν είναι υποτίθεται κράτο δικαίου, ενώ είναι αδύνατο να τα δικάζονται τέτοιοι άνθρωποι ε, και σαπίζουν στις φυλακές. Άλλοι που έχουν αθωθεί από τις κατηγορίες βλασφημίας δέχονται ε, προσβολές, ακόμα και οι δικηγόροι που είναι αρκετά θαραλέοι για να υπερασπιστούν ε, τους κατηγορούμενους κινδυνεύουν από χλοκρατία και, ε, ή και ακόμα και φόνο. αυτά επανειλημμένως τα έχουμε ακούσει και δεν έχουμε δει καμία βελτίωση. Ή και η ώρα το Πακιστάν να αγκαλιάσει τις υποχρεώσεις του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το συνταγματικό δικαίωμα που οφείλει τους πολίτες του να τους προστατεύσει. Είτε είναι χριστιανοί, μουσουλμάνοι, Ινδουιστές ή Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και δίνω το λόγο τώρα στον τελευταίο των συντακτών, τον κύριο Λέναρς. Yes, thank you, Chairman. Um, I'm... ευχαριστώ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό το ότι έχουμε τώρα την ευκαιρία να συζητάσουμε αυτό το ψήφισμα κατόπιν τη συζήτηση που έγινε στην τελευταία σύνοδο. Γιατί προβληματιζόμαστε βαθιά όσον αφορά αυτούς τους επίμαχους νόμους για τη βλασφημία του Πακιστάν. Χρησιμοποιείται η έννοια αυτή για να φημώσει τον ε, λαό και τα πράγματα γίνονται λένε και πιο δύσκολα. Έχουμε ε, διάφορες ε, κατηγορίες βάσιμες που έχουν οδηγήσει σε θανατικές καταδίκες. Τα είπαμε και για την Άζια Μπίμπη, μια χριστιανή που τα δικαστηκε σε θάνατο. Επίσης θα πρέπει τώρα να πιέσουμε, να απευθύνουμε έκκληση αρχέ αρχές του Πακιστάν να καταργήσουν αυτού τους νόμους και θα πρέπει επομένω να στείλει ένα μήνυμα αποφασιστικό η Υπηρεσία εξωτερική δράση, η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσουν ό,τι υπάρχει, ό,τι έχουμε ω μέσον για να πιέσουμε τι πακιστανικέ αρχέ να κάνουν αυτή την αλλαγή. Σα ευχαριστώ. Προχωρούμε στον κύκλο των ομιλητών εκ μέρου των πολιτικών ομάδων. Εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, το λόγο έχει ο κύριο Βόμποτα για ένα λεπτό. pane eh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καμιά φορά βλέπουμε πως ε, περνάμε εμείς ψηφίσματα για τους χριστιανούς του Σουδάν ε, και άλλους ε, που καταδικάζονται σε θάνατο. Τώρα έχουμε την Άση Μπίμπη, ε, μια γυναίκα στο Πακιστάν που επίσης καταδικάστηκε σε θάνατο με βάση αυτούς τους νόμους. Εγώ ζητώ από τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να ζητήσουν από τον πρόεδρο του Πακιστάν να δώσει χάρη στην Άζια Μπίμπη. Είναι ο απλούστερος τρόπος Ζητάω λοιπόν να επανεξετάσουμε επίσης την αναπτυξιακή βοήθεια και το προστιμησιακό καθεστώς του Πακιστάν. Γιατί ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων υποτίθεται ότι είναι όρος για αυτές τις ε, εμπορικές προτιμήσεις. Στην περίπτωση του Σουδάν έπιασε αυτή η απειλή. Σας ευχαριστώ. Δέχεστε μία μπλε κάρτα, υπάρχει ερώτηση από τον κύριο Μπασίρ για εσάς. Ναι. Κύριε Μπασίρ, κάντε την ερώτησή σας. Η ερώτησή μου είναι... Εδώ μέσα ε, συζητάμε τα δικαιώματα των χριστιανών ε, μην το κάνουμε τώρα το θέμα χριστιανοί εναντίον Ισλάμ. Ε, όλοι οι άνθρωποι είναι θύματα αυτών των νόμων. Εσείς κύριε και άλλοι αναφέρατε πολλούς χριστιανούς που διώκονται. Ε, πρέπει να ευασπιστούμε όλους τους ανθρώπους όλων των θρησκειών, όχι μόνο τους χριστιανούς. Βεβαίως. Μα βλέπουμε και βάσει τα στατιστικά στοιχεία πως ε, κυρίως οι μουσουλμάνοι ε, είναι θύματα αυτών των νόμων. Εννοείται αυτό πως ε, και για αυτούς αγωνιζόμαστε. Ευχαριστώ η κυρία Γιακονσάρη για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Πακιστανέ σημαντικό σημαντικός εταίρος. Και γι' αυτό με τους εταίρους και τους φίλους πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και άμεση. Να πούμε <coughs> άμεσα στους Πακιστανούς φίλους μας ότι πρέπει αυτές, αυτή την, αυτό το νόμο της βλασιμίας να το καταργήσετε γιατί οδηγεί στην ε, καταπίεση σε, δημόσιες, ε, σε δημόσια ταπείνωση και για τους χριστιανούς αλλά και για άλλους ε, θρησκευτικές μειονότητες και σίγουρα και τους μουσουλμάνους. Οι πακιστανικές αρχές απέτυχαν στο έργο τους, ακόμα και αν η Διεθνή κοινότητα, το ΟΙΕ, το Ευρωκοινοβούλιο αλλά και άλλοι διεθνείς οργανισμοί επανειλημμένως τόνισαν και απέτησαν την την αλλαγή πορείας. Θα πρέπει να επιτεθούμε στη πηγή, στα αίτια, από πού προέρχονται αυτές οι αδικίες και ζητούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συζητήσει ανοιχτά τα προβλήματα τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να πιέσουμε τις αρχές. Ε, Ο κύριος Μαρίνιο Πίντο ε, για ένα λεπτό. Δεν βρίσκεται στην αίθουσα ούτε και εκείνος, οπότε προχωράμε στην ε, κατάλογο ομιλητή ομιλητών με τον κύριο Κάουζο Περμόη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλουμε να υπάρχει διαχωρισμός θρησκείας από κράτους και αυτό αφορά για όλες τις θρησκείες. Όμως θα πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω σε, πέραν του να προβαίνουμε σε δηλώσεις για αυτούς τους νόμους. Ε, γι' αυτό και ευθύνουμε έκκληση το Πακιστάν να καταργήσει αυτούς τους νόμους, να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο, να συμμορφωθεί με την σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και να καταργηθεί η θανατική ποινή. Πάντως ε, αυτό το οποίο επίσης δεν βοηθάει είναι οι παρεμβάσεις της Δύσης. Είδαμε τι μας είπε το για το, για, το, ε, για το βραβείο και επίσης είπαμε τι έγινε με τα drones αλλά επίσης και για το Βελοχιστάν. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στην ε, κυρία Τζιν Λάμπερτ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να σας μιλήσω ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας ε, του Κοινοβουλίου για την Οριανατολική Ασία, εκεί που πάγεται και το Πακιστάν. Και για άλλη μια φορά σας διαβεβαιώ, συνάδελφοι, ότι η αντιπροσωπεία μας όποτε πηγαίνει εκεί ε, στις, στις ανώτατες αρχές της χώρας ε, θίγουμε αυτό το ζήτημα και αναγνωρίζεται και από πλευρά τους το ότι θα πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή όχι μόνο για τις μειοψηφίες τις εθνοτικές αλλά και για τους Πακιστανούς σε ό,τι και αν πιστεύουν δεν θα πρέπει ε, να είναι σε τέτοια θέση ούτως ώστε να ε, υπάρχουν βάσιμες αναπόδεικτες κατηγορίες ε, πρέπει πάντως η αλλαγή να γίνει αλλά όλα αυτά όποιος τα λέει εκεί βρίσκεται πραγματικά σε κίνδυνο ζωής χρειάζεται πολύ θάρρος και οπότε θα πρέπει να αλλάξει η κατάσταση στη χώρα έτσι θα έχουμε τις ε, αλλαγές που θέλουμε. Α, και πώς θα γίνει αυτό. Θα πρέπει να στηριχθεί η παιδεία. Αυτό δεν υπονομεύει το Ισλάμ, αλλά υπονομεύει αυτούς που χρησιμοποιούν το Ισλάμ για τους μικροπολιτικούς στόχους. Έχουμε μπλε κάρτες, δύο υπερωτήσεις από τον κύριο Καρίμ και από τον κύριο Τάνοκ. Δέχεστε. Δέχεστε αυτές τις δύο υπερωτήσεις, επαναλαμβάνει ο Πρόεδρος. Από τους κυρίους Καρίμ και Τάνοκ. Κύριε Καρίμ, έχετε το λόγο. Um, uh, Κυρία Λάμπερτ, είστε πρόεδρος της αντιπροσωπείας της Αρμοδίας και είπαμε ότι έχουμε πει ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν το καθεστώς λοιπόν σε σχέση με, το... με τις γενικευμένες προτιμήσεις με το σχετικό μηχανισμό και θα πρέπει να δούμε ποιος θα υποστεί τις συνέπειες ε, αν προβούμε σε τέτοια αναθεώρηση των όρων ε, εμπορίας. Πάρα πολύ πρόσφατα προέδεσαν οι αρχές ε, του Πακιστάν σε 40 συλλήψεις. Τι γίνεται με αυτές τις εξελίξεις. Συμφωνείτε μαζί μου ότι το Πακιστάν ζητεί την βοήθειά μας. αυτό είναι πιο αποτελεσματικό από το να έχουμε το να ψήσουμε μετά το άλλο. Κύριε Τάνοκ, ε, ρωτήστε, αλλά αφού απαντήσει την πρώτη ερώτηση ε, η κυρία Λάμπερτ. Παρακαλώ κύριε Τάνοκ, περιμένετε να απαντήσει η κυρία Λάμπερτ και μετά ε, ρωτήστε. Um, σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ναι, θεωρώ ότι θα πρέπει να τηρούμε το, το, ό,τι προβλέπεται όσον αφορά την εμπορική μας ε, πολιτική και γενικότερα. Θέλουμε να έχουμε μία συνεπή προσέγγιση σε όσα κάνουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικός ο μηχανισμός αυτός με τις ε, επιδόσεις τέλο πάντων, scorecard. Και θα πρέπει να σταματήσουν στο Πακιστάν να χειραγωγούν έτσι, τους νόμους και θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στο ε, κράτος αυτό να προβεί στις κατάλληλες αλλαγές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να αποχωρήσουμε από το στάνταρ ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τηρούμε, που έχουμε. Κυρία Λάμπερτ, λέει ο κύριο Στάνο, και εγώ θέλω να συμφωνήσω με τον ε, συνάδελφο Καρύμ όσον αφορά την scorecard, ε, όσον αφορά τις έρευνες, όσον αφορά τις συλλήψεις, αλλά για μα μας εσείς που τα ξέρετε καλά, ε, σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Μπασίρ προηγουμένως, ε, που είπε κάτι για την προστασία των χριστιανών και λοιπά ε, και άμα δείτε τα στατιστικά, και οι, οι ΣΥΙΤΕΣ και, και ακόμα και οι μουσουλμανικές μειονότητες θίγονται εκτός από τους χριστιανούς. Επομένως το, το θέμα είναι τι θα κάνει το Ισλάμ με τις μειονότητες. Λάμπερτ. Όχι, δεν θα θεωρήσω ότι είμαι ειδική σε αυτά, αλλά τέλος πάντων, όσον αφορά το ποιοι στοχοποιούνται από ό,τι ξέρουμε, ναι, είναι αλήθεια ότι έχουν θυγεί και πάρα πολλέ μειονότητε ε, και μουσουλμανικές. Μπορεί να θεωρήσει ότι αυτό είναι πολιτική χειραγώγηση του νόμου, πολλές φορές επίσης ε, είναι ξεκαθάριση λογαριασμών σε τοπικό επίπεδο, αλλά όταν ασχολούμαστε με αυτό το θέμα θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να το παρουσιάζουμε τα πράγματα, να μην λέμε κάτι το οποίο να εμφανίζεται ως αντιισλαμισμός, γιατί αυτό είναι νερό στο μήλο αυτών που δεν θέλουν την μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καστάλτο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι ε, όροι, ε, συναδελφοί, είναι μια έννοια πολύ σημαντική, αλλά και μια έννοια την οποία καταχρώμεθα. Το Πακιστάν είναι παράδειγμα για το πώς η συνοχή επηρεάζεται από τις διάφορες εμπορικές δράσεις. Εποφασίστηκε το, ε, το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων συν μια προτιμησιακή εμπορική πρόσβαση για χώρες για τα εμπορεύματα διαφόρων χωρών με την προϋπόθεση να κυρώσουν τη Διεθνή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πώς όλα αυτά συμβιβάζονται τώρα με το νόμο περί βλασφημίας που ορισμένες φορές οδηγούν και στην θανατική ποινή. Ε, τι είναι κρίση ε, ε, όραση της Κομισιόν δεν το είδε. Ε, είναι πράγματα αυτά που μας καθιστούν λίγο αξιόπιστους και δεν βοηθούν τους Πακιστανούς. Το να μην αγανακτούμε για όλα αυτά είναι η πραγματική βλασφημία κατά τη γνώμη μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε λάβει μια μπλε κάρτα από τον κύριο Μπασίρ. Τη δέχεστε? Κύριε Μπασίρ. Αφού ήδη είχατε μπλε κάρτα, είναι η τελευταία μπλε κάρτα που δέχομαι από εσά, κύριε Μπασίρ. Ο συνάδελφος συμφωνεί ο κύριος Κοστέλο πως ε, πολλά από τα εγκλήματα στον τρίτο κόσμο και ειδικά στο Πακιστάν οφείλονται στη φτώχεια και είναι σωστό να τιμωρούμε μια χώρα και άρα να την καταδικάζουμε ακόμη περισσότερο στη φτώχεια όταν έχει αντιμετωπίσει τόσα πράγματα είναι κρίμα να τιμωρούμε μια χώρα και έτσι να την καταδικάζουμε ακόμη περισσότερο στη φτώχεια Σας ευχαριστώ όπως ε, ανέφερα εγώ είμαι κάποιος που διαρκώς το καταγγέλλω, αλλά τι έχει να κάνει αυτό με την ανοιξή θρησκεία και την ελευθερία σκέψης. Πιστεύω ειλικρινά πω η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναπτύξει σημαντική και υγιή εμπορική και πολιτική σχέση με το Πακιστάν. Και ακριβώ γι' αυτό το λόγο ω φίλοι θα πρέπει να θυμίσουμε στου φίλου μα, ότι όπω εμεί πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο ώστε να επιτρέψουμε την ανάπτυξη στι χώρε που αυτή τη στιγμή είναι σε ανάπτυξη σε σχέση με εμά, να προσπαθήσουν να δώσουν μεγαλύτερη ελευθερία στη θρησκεία και στην σκέψη. Θα πρέπει, η προσέγγιση μας θα πρέπει να είναι περισσότερο για περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο Τζανλούκα για ένα λεπτό. Η υπόθεση του Πακιστάν είναι προφανή. Η Ευρώπη βοηθάει το Πακιστάν και το Πακιστάν καταστρέφει τι μικρομεσαίε μα επιχειρήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ιταλικό επίπεδο. Έκαψαν δύο χριστιανού και εδώ κάνουμε λε και δεν τρέχει τίποτα. Όμω μόλι ο Πούτιν πει μια κουβέντα, ε, γανακτούμε κατά του Πούτιν και τη Ρουσία. Μα είστε δειλοί, πρέπει να ξυπνήσετε. Εγώ κάνω την εξή πρόταση. Η λύση για να βελτιωθεί η Ευρώπη και να ευτυχήσει και το Πακιστάν είναι πάρτε τον Κατάινεν και τον Γιούνκερ, στείλτε τους στο Πακιστάν να μείνουν εκεί και γιατί η Ευρώπη μάλλον γιατί ο Γιούνκερ εδώ προσπαθεί να μας κοροϊδέψει λέει ότι έχει 300 δις ενώ δεν έχει παρά μόνο 20. Εδώ δεν λειτουργεί τίποτα. Ξυπνήστε πια. Πέρα από το Πακιστάν δεν λειτουργεί τίποτα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Δεν θα ε, γίνουν άλλα σχόλια. Λοιπόν, αντάκτουσον για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, το Πακιστάν είναι μία από τις πιο επικίνδυνες χώρες ε, του κόσμου για τους ε, χριστιανούς. Και τελευταία οι νόμοι αυτοί είχαν καταστροφικές συνέπειες. Μία κατηγορία για βλασιμία αρκεί για να σκοτωθεί κάποιος. Αυτό το οποίο συνέβη στο Ανατολικό Πακιστάν στις 7 Νοεμβρίου είναι ένα τραγικό παράδειγμα της ε, υπόθεσης αυτής μια κατηγορία κατά του ζεύγους Μπίμπι οδήγησε σε ε, επίθεση και τους κάψαν ζωντανούς και μια σειρά προσωπικότητων του Πακιστάν με διαβεβαίωσαν πως σέβονται τα δικαιώματα όλων αλλά πολλοί αμφιβάλλουν από αυτού Εξού και η απέτησή μου στους υπεύθυνους του Πακιστάν. Σεβαστείτε την ανεξιθρησκεία και τηρήστε τον νόμο για να μην επαναληφθούν τέτοια πράγματα. Σας ευχαριστώ κυρία Γκόμες. Όταν το 2003 έστειλε το, 2000, ε, έστειλε το Κοινοβούλιο μια αποστολή ο αποκεφαλής υποσχέθηκε αλλαγή της κατάστασης. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτές οι υποσχέσεις για να αναθεωρήσουμε, ε, για, για να επικυρώσουμε μάλλον το πακέτο γενικευμένων προτιμήσεων για το Πακιστάν. Όμως η κατάσταση επιδεινώνεται και σχεδόν καμία πρόοδος δεν έχει σημειωθεί έκτοτε. Πέρα από τη βλασφημία εμποδίζεται η ανεξιθρησκεία, καταστέλλονται οι μειονότητες, οι χριστιανικές, ε, και οι μουσουλμανικές, ε, σιτικές, οι σουνιτικές. Ε, το... Το Πακιστάν βυθίζεται και μάλιστα δίθεν η προπαγάνδα κατά των τρομοκρατικών κατακαιρματίζει την κοινωνία των πολιτών που θέλει να ζήσει σε ένα ελεύθερο και δημοκρατικό Πακιστάν. Εμείς πρέπει λοιπόν να περάσουμε ένα σαφές μήνυμα και να βοηθήσουμε τους όσους στο Πακιστάν αγωνίζονται υπέρ της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ. Δέχεστε μπλε κάρτα από πλευράς ε, του συνδέλφου Καν. Κύριε Καν. 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ερώτημα που θα ήθελα να κάνω είναι δέχεστε πως κάποιοι εδώ ζήτησαν να ανασταλεί η συμφωνία γενικού συστήματος προτιμήσεων. Εάν είναι να βοηθήσουμε τα θύματα και να υπάρξει αλλαγή, πρέπει να συνεργαστούμε με το Πακιστάν. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε να τους απειλήσουμε. Απάντηση. Κατά την άποψή μου πρέπει να καταργηθούν οι νόμοι περί βλασφημίας οι οποίοι αντιβαίνουν σε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα που ήταν προϋπόθεση για, τις, για το σύστημα προτιμήσεων Τώρα δεν ξέρω αν θα ήταν θετικό ε, αλλά πρέπει να είναι στα υπόψη αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Δεν είναι δυνατόν να υπακούει την Σαουδική Αραβία και να προωθεί τους νόμους αυτούς που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα χριστιανών και μουσουλμάνων. Σας ευχαριστώ. Μπρόνισλαβ Σκρίμπακη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, φανταστείτε να είχατε την αδερφή σας εκεί και να είχε καταδικαστεί σε θάνατο εκεί στο Πακιστάν. Ε, ε, Συμπολίτε μας είναι θύματα και φυλακίζονται εκεί. Είδατε τι γίνεται με το μίσος που υποδαβλίζεται από την ε, θρησκεία. Αυτό έγινε και με την κυρία Μπίμπη. κατηγορήθηκε, ε, αφέθηκε νηστική, χωρίς νερό, ε, ε, δάρια, όλα αυτά επί τη βάση αυτών των νόμων για τη βλασφημία. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να σώσουμε την μητέρα πέντε παιδιών στην Ανατολική Ευρώπη. Γνωρίζουμε καλά αυτές τις καταστάσεις. Τα έχουμε περάσει. Τι θα πει δίωξη βασισμένη στην θρησκεία. 25 χρόνια τότε που άλλαξε το καθεστώς είναι αλήθεια ότι η θρησκευτική ελευθερία είναι μια πολυτέλεια και στο Πακιστάν αλλά και σε άλλες χώρες δεν υπάρχει αυτή η ελευθερία. Εκφοβισμός. Αυτό είναι η ντροπή. Θα πρέπει να σταματήσουμε αυτού του είδους ε, τους πα, παράλογους νόμους. Ο πρόεδρος. Ένα λεπτό Μαρίνια Πίντα. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, καμία θρησκεία δεν μπορεί να δικαιολογήσει την βαρβαρότητα και την αγριότητα. Καμία θρησκεία δεν μπορεί να δικαιολογήσει ότι ένας οργισμένος όχλος να, να θανατώσει ένα χριστιανικό ζευγάρι ε, να τους κάψει στους φούρνους εκεί που εργαζόταν. Καμία θρησκεία δεν μπορεί να αιτιολογήσει ε, τον ε, θανάτωση του Υπουργού που ήταν χριστιανός ακριβώς και μόνο επειδή επίκριναν τον νόμο περί βλασφημίας και μίλησαν υπέρ της προστασίας των θρησκευτικών μηνοτήτων. Κανένα νόμος δεν μπορεί να αιτιολογήσει την καταδίκη σε θάνατο πάνω από χιλίων ε, ε, ανθρώπων μεταξύ αυτών και της Άζια Μπίμπι. Καμενένας νόμος δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη θανάτωση ενός δικηγόρου που υπερασπιζόταν στο δικαστήριο κάποιον που είχε κατηγορηθεί για βλασφημία. Αρκεί η βλασφημία. Χρειάζεται το Πακιστάν να μπει στην κοινότητα των πολιτισμένων κρατών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπανσίρ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, εγώ καταδικάζω εντόνως τη βία τη βία δολοφονία Σάμα και Σανμπάζερ και Πακιστανών χριστιανών από τον όχλο καθώς και τις υπόλοιπες καταχρήσεις που γίνονται στο όνομα της βλασφημίας. Αυτές οι βαρβάρες πράξεις δεν μπορούν να είναι αποδεκτές στο Ευρωκοινοβούλιο, στη διεθνή κοινότητα και το πακιστανικό έθνος. Γνωρίζω ότι το πακιστανικό έθνος βρίσκεται σε μια κατάσταση σοκ και είναι εξοργισμένο. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι αυτοί οι νόμοι υπάρχουν στο Πακιστάν από την εποχή της απεικιοκρατίας και ότι οι περισσότερες υποθέσεις υπό αυτή την νομοθεσία ήταν εναντί μουσουλμάνων. Εγώ ε, ε, έλαβα διαβεβαιώσεις από τις πακιστανικές αρχές ότι έλαβαν τα απαραίτητα βήματα ώστε να επιβεβαιώσουν πιθανές καταχρήσεις των ισχυών των νόμων. Θα πρέπει επίσης να θυμίσουμε ότι κανένας μέχρι στιγμής δεν έχει τιμωρηθεί με βάση αυτές τις νομοθεσίες. Οι υποθέσεις που στοιχειοθετούνται υπό την νομοθεσία ε, δεν υπέστησαν δικαστική κόελεγχο στα διάφορα επίπεδα κατέστη υποχρεωτικό κανένας αστυνομικός ε, να μην μπορεί να ερευνήσει τις κατηγορίες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σοπράντ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, τον Νοέμβριο του 2010 η Άζια μια χριστιανή Πακιστανή, κατεδικάστηκε στην θανατική ποινή από τις αρχές της χώρας της με το αίτιο ότι προσέβαλε τον Μοχάμετ. Έκτοτε οποιαδήποτε απόπειρα έφεση έναντι αυτής τη απόφασης απερίφθη. Ε, περιμένει στο διάδρομο του θανάτου την απόφαση του ανώτατου Πακιστανικού Δικαστηρίου που είναι το τελευταίο της ε, καταφύγει για να σώσει τη ζωή της. Ε, θα ήθελα να θυμίσω εδώ, συνάδελφοι, ότι σύμφωνα με το μαύρο βιβλίο τη συνθήκη των χριστιανών στον κόσμο, ανάμεσα σε 120 και τα 200 εκατομμύρια χριστιανών υπόκειται σε διωγμούς. Σημαίνει αυτό ότι χιλιάδες άνθρωποι κινδυνεύουν καθημερινά μόνο και μόνο επειδή πιστεύουν τον Χριστό. Ωστόσο, Ακόμα μια φορά η, η περιφέρεια ιδεολογία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, ε, καλύπτει τα πάντα και γι' αυτό και δεν πρόκειται να στηρίξω αυτό το ψήφισμα. Δεν θα στηρίξω ακόμα μια φορά το ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει μόνο στόχο να καταλύσει την κυριαρχία των κρατών ώστε να, ε, ευνοήσει τις ολιγαρχίες που εξυπηρετούν αυτές τις προθέσεις. Εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχίσει να κάνει την εκαθάριση στις Ισλαμιστικές οργανώσεις εδώ. Η Αζιαμπίπη δεν θα σωστεί από εμά, αλλά από μια Ευρώπη που θα αναλάβει και θα δεχτεί τον χριστιανικό της πολιτισμό και θα προσφέρει προστασία στους χριστιανούς στην ίδιες τους τις χώρες. Ο Πρόεδρος. Τώρα έχουμε τη διαδικασία κατσιτιάε. Δέκα συναντηθούν στο λόγο, οι περισσότεροι από του οποίου προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Πάντως, Έχω αποφασίσει, λέει ο Πρόεδρος, να δώσω το λόγο σε όλους τους συναδέλφους που έχουν ζήσει το λόγο. Αλλά παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο του ενός λεπτού, για έτσι να μπορέσετε όλοι να μιλήσετε. Ο κύριος Σόγκορ, ε, πρώτος, έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όπως συμβαίνει και με άλλες μειονότητες, έτσι και οι Βαλούχοι έχουν πληγεί. Κάτι το οποίο αποδεικνύει πως δεν μπορεί να προστατεύσει τις ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας του. Το Πακιστάν οι νόμοι περί βλασφημίας παραβιάζουν το Διεθνές Σύμφωνο Πολιτικών Δικαιωμάτων το οποίο πρέπει να τηρήσει το Πακιστάν εάν θέλει να συνεχίσει να έχει εμπορικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης πολλά κοσμικά κόμματα στο Πακιστάν έχουν ζητήσει την κατάργηση τη σχετική νομοθεσία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσέξει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Κάπου τον Νίκολα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Πακιστάν είναι η μοναδική μουσουλμανική χώρα που έχει νόμο για τη βλασφημία. Από το 1990, όταν εισήχθη αυτός ο κανόνας, γύρω στις 60 εκτελέσεις έχουν γίνει. Η βία της Σαρία δεν αγγίζει μόνο τους χριστιανούς, αλλά και άλλες μειονότητες. Σε αυτή την αίθουσα διαμαρτυρηθήκαμε κατά της απόφασης του ΙΠΑ του δικαστηρίου της ΑΚΟΡ να, την, να κυρώσει την απόφαση για τη θανάτωση της Άζια Μπίμπη όπως και για τους ε, δύο χριστιανούς που κάηκαν ζωντανοί από τον όχλο ακριβώς γιατί κατε, κατηγορήθηκαν για βλασφημία. Όμως αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει να πιέσουμε το Πακιστάν να προβεί στα απαραίτητα βήματα για να καταργήσει αυτή την νομοθεσία. Θα πρέπει να καλέσουμε την κυβέρνηση του Ισλαμαμπάτ να λάβει υπόψη το μορατόριο να, να, να προβεί μάλλον σε μορατόριο μου κατά της θανατικής ποινή. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας για να πιέσουμε την πακιστανική κυβέρνηση. Η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να, ε, να παρέμβει μέχρι ότου το Πακιστάν να σεβαστεί τις υποχρεώσεις του απέναντι στην ελευθερία έκφρασης και θρησκείας. Βαντάλεν τώρα. Κύριε Πρόεδρε, Δικαίως σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει να δοθεί προσοχή σε αυτή την νομοθεσία. Γιατί αθώα κάθεται τόσα χρόνια στο κελί η Άζια Μπίπη. Πρέπει να απελευθερωθεί και να γίνει γρήγορα η δίκη στο ανώτο δικαστήριο στην Λαχώρη. Η ο νόμος αυτός περί καλύπτει σαν ένα πέπλο φόβου ολόκληρη την πακιστανική κοινωνία. Δικαίως συζητάμε σήμερα και λέμε πως ε, το, ο νόμος αυτός παραβιάζει τις ε, διεθνείς υποχρεώσεις που έχει συνυπογράψει το Πακιστάν. Η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή, η κυρία Μάλμστρομ, πρέπει να ερευνήσουν γρήγορα το εάν ε, εκπληρώνονται υποχρέσεις που έχει αναλάβει το Πακιστάν ενώπιον μας. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε εμπορικές προτιμήσεις με αυτή την κατάσταση να επικρατεί. Σας ευχαριστώ. Η Ρασίντα Ντατή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφέρθηκαν πολλά και συμφωνώ με όσο είπαν οι συνάδελφοι με αυτό το ψήφισμα θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ξεκάθαρο ε, στήριξη στην κυρία Μπίμπη αλλά επίσης να θέλουμε έκκληση και στις αρχές ε, τη Πακιστανική να απελευθερώσει και να καταργήσει τον νόμο. Με αυτό το ψήφισμα θέλουμε να καλύψουμε όλε αυτέ τι διώξει για ένα σωρό κόσμο που δεν έκαναν τίποτα. Απλώ πιστεύουν στον Θεό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκάθαρα ε, υπεραμείνεται τη θρησκευτική ελευθερία για οποιαδήποτε θρησκεία κύριε Σόπραν, αλλά βέβαια και έχουμε και την ευθύνη να τον των χριστιανών, διότι έχουμε μια πολιτική ταυτότητα ε, και οι ρίζα μας είναι στον χριστιανισμό. Εάν δεν επεραμεινθούμε αυτά τα 150 εκατομμύρια των χριστιανών που διώκονται σε όλο τον κόσμο, ποιος θα το κάνει. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα δώσουμε το λόγο στον κύριο Μάρεκ Γιούρεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, αναφέρθηκε ε, ο κ. Φαντάλεν, ε, ο κ. Σόπρα, διότι ανέφεραν την περίπτωση της κυρίας Βίμπη. Και εγώ θα ήθελα να σας προτείνω να γίνουμε πιο ρεαλιστές, να αναλάβουμε δράση. Δεν είναι δυνατόν να βασανίζεται έτσι, δεν είναι δυνατόν να, βρίσκεται στην πτέρυγα των μελοθανάτων. Οι, οι αρχές της χώρας μου είπαν ότι ε, θέλουν να παρέμβουν. Και το ίδιο είπε και ο Δήμαρχος των Παρισιών, δηλαδή θα πρέπει να αναλάβουμε διπλωματικές ενέργειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Μογκερίνη είπε ότι εκπρόσωπος να αναλάβει τις πρωτοβουλίες αυτές. Ε, κράτη μέλη επιτόπου ε, να παρέμβουν και θα πρέπει να αποφυλακιστεί η κυρία Μπίμπη θα πρέπει να λέμε στους μουσουλμάνους ε, συνομιλητές ότι εμείς δεν διώκουμε τους μουσουλμάνους για τη θρησκεία τους και το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και από πλευρά τους. Κυρία Μαριάννα Πέτρη. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η θανατική καταδίκη της Αζία Μπίμπη πρέπει να ανατραπεί. Πρόκειται για χριστιανή, μητέρα πέντε παιδιών, και είχε συλληφθεί με την κατηγορία της λασιμίας και απαιτώ να απαιτεί ελεύθερη. Επίσης απαιτώ αυτοί που σκότωσαν τους δύο χριστιανούς, ε, το ζευγούς, Μπίμπι να συλληφθούν. Τους έκαψαν ζωντανούς. Επίσης απαιτώ να ανακληθεί ο νόμος περί βλασιμίας του Πακιστάν γιατί παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την Η γνώση είναι πως το Πακιστάν παίζει σημαντικό ρόλο στη σταθερότητα στην Νοτιοανατολική Ασία. Γι' αυτό ζητώ από τις πακιστανικές αρχές να ηγηθούν δια του παραδείγματος, ε, ενισχύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι παραβιάζοντάς τα. Τον λόγο έχει ο κύριος Καρύμ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Είμαι υπερήφανος για το ότι γίνεται αυτή η συζήτηση σήμερα εδώ. Προχτές ο Πάπας μίλησε εδώ και ξεκαθάρισε πως η Ευρώπη δεν τηρεί τις αξίες της, χάνουμε τον δρόμο μας. Και αυτό βλέπω σήμερα εδώ. Πολλοί από τους συνάδελφους μας ίσως δεν γνωρίζουν, αλλά το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχουν παίξει τεράστιο ρόλο στην απελευθέρωση ενός Ευρωπαίου πολίτη που ανέμενε εκτέλεση στο Πακιστάν. Στο Αυτό το καταφέραμε πριν από λίγα χρόνια. Δεν υπάρχει λόγος ο διάλογος μας να μην μας επιτρέψει να ε, έχουμε ξανά τέτοια επικοδομητικά αποτελέσματα. Για την Κομισιόν να πω το εξής. Ναι, ακούσαμε διάφορα πράγματα ε, για τις εμπορικές μας σχέσεις με το Πακιστάν. Μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις ε, δώσαμε το πρωτομησιακό καθεστώς στο Πακιστάν και υπάρχει ένας πίνακας βαθμολογίας. Ας τον εφαρμόσουμε. Πρέπει όλοι εδώ πέρα να συνεργαστούμε με το Πακιστάν για να επιτύχουμε τον στόχο μας να σώσουμε ζωές. Ευχαριστώ. Η κυρία Σουίτσα. Καμία θρησκεία δεν μπορεί να δικαιολογήσει και να στηρίξει τέτοιου είδους πράξεις. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ό,τι μέσα έχουμε στην ε, διάθεσή μας. 150 είναι τα εκατομμύρια των χριστιανών που διώκονται σε όλο τον κόσμο και έχουμε και τον νόμο για τη βλασφημία του Πακιστάν που είναι κάτι το κατασταλτικό, κάτι το απαράδεκτο να μην μείνουμε σταυρωμένα χέρια. Θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη ότι εδώ δολοφονήθηκαν αυτοί οι δύο Πακιστανοί οι χριστιανοί, είδα από την Ασιαβή που βρίσκεται τώρα στα, στα πρόθεση ανεδικής ε, ποινής, της, ε, της εκτέλεσης μάλλον, και αυτό γιατί άσκησε θεμελιώδη δικαιώματα. Άρα θα πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα. Δεν είμαι βέβαιη ότι θα φέρει ε, κάποια αποτελέσματα. Κυρία Στυλιανίδη, η αναπτυξιακή βοήθεια στέλνεται στο Πακιστάν. Οπότε θα πρέπει να θέσουμε κάποια καινούργια πλαίσια για τη συνέχιση αυτής της ε, βοήθειας. Να υπάρξει κάποια επικοδομητική πρόταση. Ευχαριστώ κύριε Αλεγκρίπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στο όνομα των, αξιών, των καθολικών αξιών που είναι ιδρυτικές όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ελευθερία έκφρασης, σκέψης, συνείδησης, ε, θρησκείας, ε, η θρησκευτική ανοχή που κάνουμε έκκληση προς τις αρχές του Πακιστάν να καταργήσουν τους νόμους περί βλασφημίας. Ε, το ίδιο το Σύνταγμα του Πακιστάν, θυμίζω, εγγυάται τα δικαιώματα των μειονοτήτων και το ανεξιθρησκείας, το δικαίωμα κάθε μειονότητας και κάθε θρησκευτική μειονότητα. Εμεί ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πετήσουμε από τον Παγκεστάνο εταίρο μα να σεβαστεί τι δεσμεύσει του και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί όμω να κρυβόμαστε ε, πρόκειται για τους χριστιανούς. Οι χριστιανοί είναι αυτοί που διώκονται περισσότερο σε ολόκληρο τον κόσμο. Η υπόθεση της Άζια Μπιμπή, της ε, νέας αυτής γυναίκας ε, που πρέπει να βγει από τον διάδρομο του θανάτου, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ελευθερώσουμε την Άζια Μπιμπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τηλιανίδης. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, εκ μέρους της κυρίας Τερίγα Μογγερίνη της υπάτησης εκπροσώπου θέλουμε να χαιρετήσουμε την έγκριση αυτού του ψηφίσματος για τον ε, νόμο περί βλασφημίας ή τους νόμους περί βλασφημίας γιατί υπάρχουν κάποιες ε, καθημερινές γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ελευθερία στην πίστη και ε, την έκφραση και ε, την θρησκευτική πίστη. Οπότε αυτού του είδους ε, οι νόμοι έχουν πάρα πολύ βλαπτικά αποτελέσματα και απαγορευτικά όσον αφορά την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων. Οπότε από πλευρά ε, γενική αρχή εμεί καταδικάζουμε αυτού του είδου την ποινικοποίηση των θρησκευτικών πεπιθήσεων γιατί αυτή οι νόμοι περί βλασφημίας χρησιμοποιούνται ούτως ώστε να ξεκαθαρίζονται λογαριασμοί και ε, χρησιμοποιούνται στις ε, αντιπαλότητες ε, διαφορετικών θρησκευτικών δογμάτων εκεί. Οπότε προβληματίζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό όχι μόνο γιατί αυτές οι κατηγορίες οδηγούνται σε θανατική ποινή. Αλλά τον Ιούνιο αρχίσαμε ένα διάλογο με το Πακιστάν και συζητήσαμε τους νόμους περί βλασφημίας. Οπότε υπενθυμίσαμε ότι θα πρέπει το Πακιστάν να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει όσον αφορά τα δημοκρατικά θεμελιώδη δικαιώματα που περιέχουν βέβαια και την ελευθερία τη πίστης. Ε, έγινε αυτή η επίσκεψη επίση τον Οκτώβριο στο Πακιστάν, τον Οκτώβριο του 2014 του κυρίου Λαμπρινίδη ε, του εκπροσώπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οπότε και ο κ. Λαμπρινίδη ε, έθιξε συγκεκριμένα αυτού του στην ε, κατάχρηση του να επικαλούνται του νόμου Ευρωσημίας για αυτού του σκοπού. Επίση, είπε ότι προβληματιζόμαστε πάρα πολύ σοβαρά όσον αφορά την απόφαση του Ανατολικού Δικαστηρίου να επικυρώσει την καταδίκη τη κυρία Αζιαβίβη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ζήτημα οι, οι νόμοι περί βλασφημίας ε, στην ε, πακιστανική κοινωνία. Το μήνυμα μας προς τους αρχηγούς της χώρας, τους ηγέτες της χώρας, είναι ότι θα πρέπει να βρεθεί το θάρρος του, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και ότι οι απειλές ε, να σταματήσουν κατά, τους, ε, κατά όσων ασχολούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, κατά των δικηγόρων, κατά των δικαστών, όλων ασχολούνται με το πρόβλημα αυτό, γιατί έχουμε ακόμα και ανθρωποκτονία στις βάρες αυτών των προσώπων και θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο το ότι οποιοδήποτε είδους ατιμορρησία για τέτοια εγκλήματα ε, αποτελεί υπονόμευση του, της τάξη τάξης και του κράτους του δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ευκαιρία παρουσιάζεται ούτως ώστε να φύγει αυτό το ζήτημα προς ε, τους πακιστανούς συνομιλητές μας. Οπότε το σύστημα γενικών προτιμήσεων ε, Plus ε, αποτελεί ένα σοβαρό σημείο για τις σχέσεις μας με τη χώρα αυτή και το, αυτό το GSP Plus είναι ένα πλαίσιο το οποίο μας καθορίζει το πώς θα εφαρμόσουμε τις διεθνείς ε, ε, συμφωνίες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργατικά δικαιώματα, το τα δικαιώματα, τα, τις υποχρεώσεις και δικαιώματα των περιβάλλων. Και ιδίω ξέρετε, η αντιπροσωπεία μας στο Ισλαμαμπάντ πρόκειται να συνεχίσει να παρακολουθεί τις ε, εξελίξεις για την υπόθεση Αμπίμπη και επίσης θα συνεχίσει τις προσπάθειες ούτω ώστε να ανατραπεί η απόφαση της καταδίκης και να αποφυλακιστεί. Και με κάθε ευκαιρία θα συνεχίσουμε αυτή την υπόθεση ε, να την συζητούμε με τους Πακιστανούς συνομιλητές όπως και γενικότερα το θέμα των νόμων της έλαβα ε, υπόψη το πόσο ενδιαφέρεστε για το πρόβλημα αυτό και σας διαβεβαιώνω η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί και πρόκειται να συνεχίσει να συνομιλεί με το Πακιστάν και όσο με ανθρώπινα δικαιώματα και όσο εμπλεκομένους και πρόκειται να έχουμε την επίσκεψη στην Ευρώπη του Προέδρου της Πακιστανικής Γερουσίας. Θα γίνει αρχάς του 2015. Αυτό θα είναι μια ευκαιρία τόσο ώστε να ε, συζητηθεί το ζήτημα. Ευχαριστώ. Thank you, Commissioner. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, λέει ο Πρόεδρος. Έχω επίσης λάβει έξι προτάσεις ψηφισμάτων. Η ψηφοφορία για αυτή τη συζήτηση θα γίνει στις 12 η ώρα. Πάμε όμως τώρα στο επόμενο θέμα της ευρεσίας διατάξεως. Πρόκειται για την υπόθεση του κατηγορουμένου για εγκλήματα πολέμου Σέσελη. Και θα δώσουμε τον λόγο στον κύριο Ιγνάτζιο Κοράου για ένα